Συνάδελφοι, καθίστε. Είμαι η Ρίνα Μακέβαν, είμαι πρόεδρο τη Επιτροπή Ανάπτυξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλου του συναδέλφους από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και τον συμπρόεδρο, τη συμπρόεδρο, την κυρία Κίνγκα Γκάρ, πρώτη αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Σα ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα. Καλώ ορίσατε στην Επιτροπή μα. Θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα. Ένα το οποίο σχεδόν καθημερινά προβάλλεται στα μέσα ενημέρωση. Όλοι ακούμε λοιπόν στον τύπο τα θλιβερά περιστατικά με του ανθρώπου που προσπαθούν να διαφύγουν, να ξεφύγουν στο Μεσόγειο από καταστάσεις ε, που απειλούν τη ζωή τους και αυτό φυσικά απασχολεί και εμάς και τις περιφερειές μας. Άρα το αντικείμενο της σημερινής σα είναι πολύ ευαίσθητο, έχει να κάνει με τις εξωτερικές και ιστορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία, ανάπτυξη, ανθρωπιστική βοήθεια και θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν. Ανάπτυξη της ε, μετανάστευση είναι τομέας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών. Φυσικά όμως μία από τις βασικές αρχές της ε, πολιτικής ε, ανάπτυξης είναι να υπάρχει συνέπεια, συνοχή και για να υπάρχει μια σαφής πολιτική, μια πολιτική η οποία θα έχει αποτελέσματα για όσους αντιμετωπίζουν την σύγκρουση, την ακραία φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ανάπτυξη μια πολιτικής η οποία θα είναι αποδεκτή και στις δικές μας χώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο και γι' αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα τη σημερινή συνεδρίαση και ελπίζω ότι οι ομιλητές ε, όχι μόνο θα αναλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά θα μας ε, κάνουν και κάποιες προτάσεις για επίλυση των ζητημάτων. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σύνθετη και πολύπλοκη αυτή η συζήτηση. Ξέρουμε ότι στη δική μου χώρα όταν ο κόσμος λέει ότι δεν θέλουμε να αποτελούμε πυρήνα έλξης και να ε, διατρέχει ο κόσμος κίνδυνο για να έρθει στην Ευρώπη. Σε πολλές χώρες ασφαλώς τύφεται το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και ελπίζω λοιπόν να μας ε, διαφωτίσουν, να δώσουν κάποιες λύσεις οι ομιλητές. Έχουμε λοιπόν τέσσερις εξαίρετους ομιλητές μαζί μας σήμερα. Ο κ. Αμπρόση, Περιφερειακός Διευθυντής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ιστορική Οργάνωση, για την Μετανάστευση, η κυρία Ασπασία Παπαδοπούλου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, προσφύγων, τον πρεσβευτή της Αφρικανικής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Παντέο, και αυτός από αριστερά μου κάθεται, και στα δεξιά μου τον κύριο Ρόιτερ, Γενικό Διευθυντή του Σολιντάρ. Θα ήθελα εξ ονόματος και των δύο επιτροπών να σας καλωσορίσω εδώ σήμερα και προσβλέπω να ακούσω τα όσα έχετε να μας πείτε. Όπως βλέπετε είναι πολύ άριθμη η προσέλευση, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά θα πρέπει να έχει μια σαφή πολιτική στα θέματα αυτά. Κυρία Γκάλ, σας δίνω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μακέβαν. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία για κοινή ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Απασχόλησης είναι κάτι το πολύ ευπρόσδεκτο και πιστεύω ότι υπάρχει ένας κοινό ε, μέσα αρμοδιοτήτων με την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Το 2015 στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα εξετάσουμε σε μια έκθεση την ε, ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση, συνολική προσέγγιση στη μετανάστευση και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο και σίγουρα η σημερινή ακρόαση θα αποτελέσει μια περίσταση προστιθέμενης αξίας. Θα ήθελα λοιπόν να κοιτάξουμε τώρα το τι έχουμε να πούμε για τους ομιλητές. Θα ακούσουμε λοιπόν καταρχάς τον κύριο Αμπρόση, ο οποίο είναι περιφερειακός διευθυντή τη ε, Διεθνού Οργάνωσης για τη Μετανάστευση. Μου ζητήθηκε να ζητήσω από όλου του συμμελητές να τηρήσουν το χρονικό όριο των 8 λεπτών. Κύριε Αμπρόση, έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιες πτυχές που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη συζήτηση για την μετανάστευση και την ανάπτυξη, γιατί ασφαλώς έχουμε και περιορισμένο χρονικό όριο για την παρέμβασή μας. Θα ήταν λοιπόν σημαντικό να επικεντρωθούμε στα θέματα που θεωρούμε προτεραιότητες. Να ξεκινήσω λοιπόν ανα... λύοντας και διαψεύδοντας κάποιους μύθους σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Πρώτος μύθος. Η ίδια η ιδέα της μετανάστευσης και της μεταναστευτικής πολιτικής. Συχνά έχουμε την τάση να θέτουμε το θέμα της μετανάστευσης, σε θέματα ελέγχου, συνοριοφυλακής, ε, θεωρήσεων. Αλλά η μεταναστευτική πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στον έλεγχο του ποιος μπαίνει στον χώρο, στην επικράτειά μας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει και το κατά πόσον ε, αξιοποιούμε τα άτομα τα οποία έρχονται στην επικράτειά μας. Μια μετατροπή δηλαδή της τάσης μας να μην ελέγχουμε τόσο να μην εστιαζόμαστε τόσο πολύ στον έλεγχο όσο στην βέλτιστη αξιοποίηση. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί μια βασική αρχή. Δεύτερο μύθο που θα ήθελα να καταρρύψω. Συχνά, όταν μιλάμε για τη μετανάστευση και την ε, ανάπτυξη, πιστεύουμε ότι βελτιώνοντα την κατάσταση σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό καθεστώ τη χώρα προέλευση, αυτόματα μειώνουμε ή αποτρέπουμε τα μεταναστευτικά κίνημα, ε, τις μεταναστευτικές ροές. Αυτό δεν ισχύει απαραίτητα, ξέρετε. Καταρχάς, ε, η ίδια ιστορία το καταδεικνύει αυτό. Επίσης, δεν είναι σωστό αυτό ως αρχή. Το θέμα δεν είναι να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, η κινητικότητα εν γέννη, αλλά να τύχουν μια διαχείριση ε, προκειμένου να είναι επωφελείς αυτές οι ροές. Επίσης, η επιτεία η ίδια μας δείχνει ότι η μετανάστευση δεν γίνεται μόνο από πλευρά των υποαναπτυσσόμενων χωρών, υποαναπτυγμένων χωρών. Αντιθέτω, ε, η μετανάστευση γενικά ξεκινά στο σημείο της ε, καμπή, όπου υπάρχει ανάπτυξη και υπάρχει διάθεση από πλευρά του κόσμου να βελτιώσει τις ε, συνθήκε διαβίωση του Και νομίζω ότι αυτή η αίθουσα αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγμα. Οι πιο πολλοί εξήμων ε, ζούμε και εργαζόμαστε σε μια διαφορετική χώρα από αυτή που γεννηθήκαμε. Είμαστε τμήμα τη κινητικότητα, των ροών κινητικότητα ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά δεν είναι ούτε η πείνα, ούτε η απόλυτη ένδια και η ανάγκη αυτή που μας έσπρωξε να κινηθούμε και να μετακινηθούμε στην προσωπική μας ζωή σήμερα. Πρόκειται για να διαφορετικό είδος αναγκών και ιδεολογίας. Τρίτος μύθος που είναι σημαντικό να καταρρύψουμε. Όταν μιλάμε για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη, δεν μιλάμε μόνο για την ανάπτυξη του νότου, του νότιου τμήματος του κόσμου. Δεν μιλάμε μόνο για την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης και διαμετακόμισης. Δεν μιλάμε μόνο για την ανάγκη αξιοποίησης μετανάστευσης ως θετικό φορέα, αλλά και για την ανάγκη υποστήριξης και βιώσιμης μάλιστα υποστήριξης του βορρά, του άλλου τμήματος, του άλλου ημισφαιρίου. Για την αξιοποίηση λοιπόν της μετανάστευσης, για να διασφαλίσουμε και την διατήρηση του δικού μας επίπεδου και τη βελτίωση ενδεχομένω του δικού μας βιωτικού επίπεδου. Η μετανάστευση και η ανάπτυξη, όπως είπατε, αποτελούν ε, ένα περίπλοκο σύνολο συνθήκων. Είναι λίγο σαν τις τελίτσες που παίζαμε όταν ήμασταν μικροί. Στην αρχή δεν έβγαζε νόημα η εικόνα και από ένα σημείο και πέρα Όσο προχωρούσε το παιχνίδι, η εικόνα γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρη και βλέπαμε την εικόνα που έπρεπε να δούμε. Άρα, ποιες είναι οι τελίτσε που θα πρέπει να συνδέσουμε εδώ όταν μιλάμε για την ανάπτυξη και την μετανάστευση. Πολλέ και δύσκολε. Και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο πολύ σένθατη είναι αυτή η εικόνα και αυτή η σύνδεσμη, γιατί αν κατανοήσουμε το σύνθετο, το πολυσύνθετο του θέματος, αυτό θα μας κάνει να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται μια τέτοια αναλογή πολιτική. Επίσης, οι τελείες αυτές επηρεάζουν οι μεν της δε. Δεν επηρεάζει μόνο η μετανάστευση την ανάπτυξη, αλλά και η ανάπτυξη τη μετανάστευση. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν πόσο πολυσύνθετο είναι το θέμα αυτό, για να κατανοήσουμε πώς επηρεάζει η μεταναστευτική πολιτική την αγορά εργασίας, την ε, πολιτική απασχόλησης, πώς ε, επηρεάζεται και επηρεάζει την εμπορική πολιτική, την περιβαλλοντική πολιτική. Και αυτό είναι μόνο μια σχηματική αποτύπωση, χωρίς καν να επισέλθουμε στον τομέα της παιδείας, της υγείας και του καθεξής. Τώρα βέβαια ασφαλώς βρισκόμαστε σε μια ιστορική συγκυρία όπου έχει έρθει η στιγμή στο διεθνές προσκήνιο με την ε, ατζέντα μετά του 2015 και ορίζοντα του στόχου τη επόμενη 15 ετία σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική πολιτική. Τώρα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να επανεξετάσουμε κάποιε από αυτέ τι διασυνδέσει, τι αλληλουχίε, κάποιε από τι πολιτικέ που ακολουθήθηκαν έω τώρα στη συζήτηση και στην εργασία κυρίως για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Ασφαλώς αναγνωρίζουμε ότι η μετανάστευση είναι σημαντική για τους τρεις πυλώνες που έχουν τεθεί για την ατζέντα μετά το 2015, οικονομικός πυλώνας, ε, κοινωνικός πυλώνας και περιβαλλοντικός πυλώνας, πιστεύουμε ότι κάποια συγκεκριμένα ζητήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και πάντα θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και να τα έχουμε υπόψη μας και στις συζητήσεις γιατί η επιτυχία ή η αποτυχία μας θα κρυθεί από αυτό. Ένα βασικό λοιπόν στοιχείο που θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε όλες τις συζητήσεις για την πολιτική, για την ανάπτυξη και την ε, μετανάστευση είναι το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθούν αυτές οι πολιτικές. Αυτό που συνήθως αποκαλείται ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον εξή πολύ απλό λόγο. Συχνά σήμερα σε πολλά τμήματα του κόσμου οι μετανάστες αυτοί που πλήττονται και πληρώνουν το μεγαλύτερο κοινωνικό και οικονομικό τίμημα ζουν και εργάζονται σε περιβάλλοντα μη ασφαλή. Δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υποδομές, σε βασικές υπηρεσίες, είτε πρόκειται για υγεία, είτε πρόκειται για λοιπές κοινοφελεί υπηρεσίες και συχνά ακριβώς εξαιτία της θέσης τους είναι εκτεθειμένοι σε περαιτέρω διακριτικές μεταχειρήσεις, ανισότητες και ασφαλώς το να εργάζεται κανείς σε ένα τέτοιο αβέβαιο, ασφαλές περιβάλλον σε ό,τι αφορά τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα του ατόμου δεν βοηθάει την καλύτερη αξιοποίηση της συμβολής των μεταναστών. Και στην κοινωνία προέλευσης και στην κοινωνία που ζουν. Η αντιμετώπιση λοιπόν όλων των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το σωστό πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για του μετανάστες αποτελεί το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για να μπορούν οι μετανάστες να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη χώρα του αλλά και τη χώρα υποδοχή. Το θέμα των δικαιωμάτων όμω, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών σήμερα ισχύει ίσως και ακόμα περισσότερο στο, το, αυτό που αναφέρεται ως ανθρωπιστική μετανάστευση ή καταναγκαστική μετανάστευση. Σήμερα έχουμε μια σειρά μεταναστών εκτοπισμένων σε όλο τον κόσμο που αναγκάζονται να φύγουν λόγω έκτακτης ανάγκης. Έχουμε μάλιστα το μεγαλύτερο κύμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Προφανώς, αυτό δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα, δεν είναι μόνο θέμα ανθρωπιστικής αντίδρασης. Πρόκειται για ένα μεγάλο εμπόδιο για την ανάπτυξη σε μεγάλα τμήματα του κόσμου. Όχι μόνο επειδή υπάρχουν προβλήματα υποδομής, μετά από φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί λοιπά. Δεν πρόκειται μόνο για θέμα ανοικοδόμησης, πρόκειται για μια απώλεια ανθρωπίνου δυναμικού. Γιατί τα προβλήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται σωστά. Σκεφτείτε λοιπόν τι απώλειες ανθρωπίνου, απώλεια ανθρωπίνου δυναμικού έχουμε στη Συρία σήμερα. Μια γενιά η οποία χάνεται. Και πώς θα είναι η κατάσταση στο μέλλον για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και όλης της περιοχής και της περιφέρειας. Αυτό αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα. Έχουμε πολλά πολλά ακόμα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση της αντίδρασής μας σε, ανθρώπινη κρίση, σε ανθρώπινες κρίσεις. Θα πρέπει να, έχει, να υπάρχει ένας σύνδεσμος στις πολιτικές που δεν σχετίζονται απαραίτητα με την ε, πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε πρόκειται για την ανάπτυξη, είτε πρόκειται για την απασχόληση, για την εκπαίδευση, για την υγεία και θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ πιο συνεκτική προσέγγιση και ανταπόκριση στα προβλήματα αυτά. Αυτό ασφαλώς ε, ισχύει και για τον αντίκτυπο που έχει μετανάστευση στην περιβαλλοντική πολιτική. και το αντίκτυπο της περιβαλλοντικής πολιτικής στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στην μετανάστευση σε ό,τι αφορά παράγοντες ανθεκτικότητας, για την ε, περιορισμό της αλλίωσης του περιβάλλοντος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις η περιβαλλοντική διάβρωση πλήττει μεγάλα τμήματα του κόσμου και επίσης ε, να χρησιμοποιηθεί μετανάστευση για την αύξηση και την τόνωση της ανθεκτικότητας ολόκληρων κοινοτήτων ένας παράγοντας που επηρεάζει την καθημερινή ζωή. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν και η... τα περιβαλλοντικά φαινόμενα πλήττουν όλο τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε μεγαλύτερη τόλμη στην ανταπόκριση μας στα φαινόμενα αυτά. Αυτό που προσπαθώ να πω δεν είναι μόνο πόσο πολυσύνθετη είναι αυτή η σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και των άλλων πολιτικών, αλλά και πόσο σημαντική είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη και τις δύο πτυχές του φαινομένου, αν θέλουμε να καταλάβουμε τις διαφορές των πολιτικών που εφαρμόζουμε. Και επειδή μιλήσατε για λύσεις, αν είχα λύσεις για τα προβλήματα αυτά θα ήμουν αλλού φυσικά τώρα, δυστυχώς δεν έχω απαντήσεις, τουλάχιστον όχι όλες τις απαντήσεις, ένα τμήμα όμως της απάντησης, το οποίο θα ήθελα να σας δώσω. Ένα και μόνο, γιατί ακούμε ξανά και ξανά στον τύπο στις συζητήσεις πόσο σημαντικό είναι το θέμα της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Χώρα προέλευσης, χώρα υποδοχής. Ασφαλώς αυτό αποτελεί ένα βασικό παράγοντα γιατί η μετανάστευση είναι διαεθνικό, διασυνοριακό ζήτημα. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μία μόνο χώρα από μένα της. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εξορισμού προαπαιτεί συνεργασία μεταξύ χωρών. Αυτή η κινητικότητα περιέχει τη μεταφορά από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο. Άρα χρειάζεται σίγουρα συνεργασία. Το θέμα όμως είναι πώς θα πλαισιωθεί αυτή η συνεργασία μεταξύ της χώρας υποδοχής, της χώρας προέλευσης και της χώρας διαμετακόμισης. Εδώ είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η αναπτυξιακή πτυχή δεν έχει να κάνει μόνο με τη χώρα διέλευση και προέλευση, αλλά και με τη χώρα υποδοχής. Χρειάζεται λοιπόν πλήρης πολιτική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, όπως το συζητήσαμε και στο τελευταίο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Και εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Γκάλ. Θα δώσω το λόγο στο κύριο Βραντέο, μόνιμο εκπρόσωπο της Αφρικανικής Ένωσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ στις Βρυξέλλες. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε ποιες είναι οι δικές του απόψεις, από αφρικανικής άποψης. Πείτε μας και δύο κουβέντες για την ε, διαδικασία και την πρωτοβουλία για το κέρας της Αφρικής. you very Ευχαριστώ πολύ, Συμπρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνεισφέρω στην ανταλλαγή απόψεων σήμερα το πρωί. Όντως η μετανάστευση ανησυχεί όλο και περισσότερο την Ευρώπη κυρίως και σε κάποιο βαθμό και την Αφρική. Θα ήθελα επίσης να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις και σχόλια. Για τους διάφορους ε, τρόπους που λαμβάνει και μορφές η μετανάστευση, ιδιαίτερα η ενδοπεριφερειακή, ενδοπεριφερειακή και διεθνής. Το είπε και ο προλαλής σας. Η μετανάστευση θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο. Μετά το 2015, που τώρα ε, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης ε, το πρόγραμμα, υπάρχει και η ατζέντα της Αφρικής για το 2063, και ε, στο πλαίσιο της ε, σχέσης ε, και συνεργασίας και εταιρικής σχέσης Αφρικής-Ευρώπης και καθώς επίσης και στο ρόλο που θα διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το 11 πλέον, και πώς θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη. Υπάρχει ρόλος εκεί για τον ιδιωτικό τομέα, με ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κτλ. γνωρίζουμε τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη μετανάστευση, που είναι είτε προσέλκυση είτε όθηση από τις χώρες προέλευσης. Γνωρίζουμε την οξύτητα που έχουν προσλάβει οι διεθνείς ε, εγκληματικές δραστηριότητες με τράφικινγκ, με λαθρεμπόριο, ακόμα και ανηλίκων. Με αυτή την εκμετάλλευση και την επικίνδυνη έκθεση των ε, μεταναστών ε, στα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα. Δυστυχώς το κοινό έχει πάντα αρνητική εικόνα της μετανάστευσης. Σκέφτεται πάντα την παράτυπη μετανάστευση. Ενώ υπάρχουν χιλιάδες πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν από την Αφρική ή ε, από τη Μέση Ανατολή, να περάσουν τη Μεσόγειο και να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτό διαμορφώνει την κοινή γνώμη. Η εκλογή σας αρχίζουν να φοβούνται. Αν ε, κυριαρχία φρουρίου, να τους αφήσουμε απ' έξω γιατί έχουν έρθει και προσπαθούν να μας αλώσουν, να αποσταθεροποιήσουν ε, τον άνετο και ασφαλή τρόπο ζωή μας, ζωής μας, ε, τότε αυτό γιατί ισχύει σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσαρκώνεται στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν οι πολίτες και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό. Τους εκπροσώπους τους που φροντίζουν τα συμφέροντά τους και ποιους ψηφίζουν. Και δυστυχώς όλο και περισσότερο στα κράτη-μέλη της Ένωσης κυριαρχεί είναι από τα βασικά θέματα η μετανάστευση. Και τα μανιφέστα των πολιτικών κομμάτων για να κερδίσουν εκλογές ε, η πλειοψηφία θα πρέπει να έχουν ε, μια αναφορά στην μετανάστευση έτσι ώστε οι κυβερνήσεις να παραμείνουν ή να φτάσουν κάποια κόμματα στην κυβέρνηση. Επίσης, είναι ενοχλητική αύξηση κρουσμάτων, ρατσισμού και ξενοφοβίας. Όλα αυτά πώς τα αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως και προφανώς δεν μπορούμε να εμποδίσουμε κανέναν να μεταναστεύει ανέκαθεν υπήρχε στο παρελθόν μετανάστευση σε διάφορες συνθήκες και δεν πρόκειται να καταργηθεί. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε κανέναν να κινείται. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις μεταναστευτικές ροές έτσι ώστε να επωφεληθούν όλοι. Και μιλώ εδώ για τρεις πλευρές. Ε, κερδίζει η χώρα προέλευσης, κερδίζει η χώρα προορισμού, κερδίζει ο ίδιος ο μετανάστης έχουμε διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις που μας δεσμεύουν και θα πρέπει να τηρούμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών είναι κρίσιμος παράγων για μας και θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ευάλωτοι, που είναι σε κίνδυνο και για τους εαυτούς τους και για τις οικογένειές τους. Παρόλα αυτά έχουν την προσδοκία να βρουν μια καλύτερη ζωή, την οποία επιδιώκουν. Δεν επιδιώκουν να είναι βάρος στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης καμίας χώρας. Θέλουν να πάνε στη χώρα αυτή και να είναι πολύτιμα μέλη της κοινωνίας, να βρουν δουλειά, να κανονίσουν τη ζωή τους κτλ. Μια φυσιολογική ζωή. Βλέπουμε και ε, κάποια δόση υποκρισίας όταν ομιλούμε για μετανάστες στην οικονομία μας βλέπουμε ποια είναι η δημογραφική κατάσταση και η πολιτική και η κοινωνική. Αυτό απαιτεί ένα κυνήγι κεφαλών εντό εισαγωγικών. Στοχεύουμε συγκεκριμένε κατηγορίες που μας χρειάζονται και με πολύ μεγάλη προθυμία πηγαίνουμε και τους βρίσκουμε. Ποιου προσελκύουμε όμως ως μετανάστες. Θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποια προσόντα, δεξιότητες, μόρφωση για να μπορούν να ενταχθούν στις ανάγκες που έχουμε εμείς ε, σε ένα μεγάλο ρυθμιστικό σχέδιο για την ε, απασχόληση, τη μετανάστευση. Όταν οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή ειδίκευση, ε, που είναι σε άλλη ηλικιακή κατηγορία, που θα μπορούσε η αγορά να τους απορροφήσει, δείχνουμε πολύ μεγάλη προσοχή για να μην πω διστακτικότητα Ακόμα και οι διαδικασίες για τη χορήγηση θεώρησης που θεσπίζουμε καθιστούν αδύνατο σχεδόν ε, για τους ανθρώπους αυτούς να έρθουν ως κανονικοί μετανάστες, νόμιμοι. Θα πρέπει και αυτό να το κοιτάξουμε ενδεχομένω και πώς εφαρμόζουμε και ποιες πολιτικές θα εφαρμόσουμε που να είναι επωφελής. επωφελείς. Win-win. Αυτό ασφαλώς θα γίνει με διεύρυνση και ευάθυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Και έτσι θα αυξηθεί και η κινητικότητα των εργαζομένων. Has Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώνεται και αυξάνει τα μέλη της, προσπάθησε να εμβαθύνει και την ολοκλήρωσή της. Και είδαμε πώς μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα εντός των κρατών μελών από την κινητικότητα των εργαζομένων. Πολλό δε μάλλον για ε, ανθρώπους που έρχονται στην Ένωση εκτός αυτής. Αυτό που χρειάζεται ειλικρινά είναι να φύγουμε από τα λόγια και να περάσουμε στα έργα. Έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα πάρα πολύ καιρό. δεν μπορεί να είναι στα τυφλά η πολιτική μας ή στο πόδι. Χρειάζεται δέσμευση πολιτική για να υπάρξει ουσία σε οποιαδήποτε συμφωνία και πλαίσια πολιτικής καταλήξουμε. Στο διάλογο λοιπόν για τη μεταναστευτική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής έχουμε έξι θεματικές ενότητες. Δουλεμπόριο μεταναστών, παράτυπη μετανάστευση, εμβάσματα, ε, κινητικότητα εργαζομένων, διασπορά και διεθνής προστασία. Υπάρχει πρωτοβουλία με το κέρας της Αφρικής για το τράφικινγκ και το δουλεμπόριο. Το Οκτώβριο του 2014 κίνησε αυτή η προσπάθεια στη Χαρτούμ. Έχουμε και ένα κοινό πρόγραμμα που ενέκριναν το Ιανουάριο του 2015 τα κράτη-μέλη μας, πριν από δύο μήνες μόλις. Η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κέρατος της Αφρικής ληφθεί αμέσως μετά τα πολύ τραγικά τεκτενόμετα στη Λαμπετούζα, αλλά χρειάστηκαν 18 μήνες περίπου για να γίνει η πρώτη συμβουλευτική διάσκεψη και στη συνέχεια η πρώτη περιφερειακή υπουργική διάσκεψη τον Οκτώβριο του 2014 για το δουλεμπόριο και τη διακίνηση ανθρώπων. Ποιο στόχο έχει αυτή η πρωτοβουλία να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της περιοχής εκεί για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του τράφικινγκ και της διακίνησης ανθρώπων από ε, το της Αφρικής. Οι περισσότεροι από τους μισούς Αφρικανούς ε, που ζητούν καλύτερη ε, ζωή, καλύτερη εργασία γίνεται στο εσωτερικό της Αφρικής. Και ε, θα αυξηθεί ο αριθμός των Αφρικανών που θα χρησιμοποιούν επικίνδυνους και αβέβαιους διάβλους. Γι' αυτό ε, είναι ένα πρόβλημα για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς της Αφρικής για αηφόρο και βιώσιμη την περασμένη εβδομάδα μια στρογγυλή τράπεζα στο Κικάλι, στη Ρουάντα, συμφώνησε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων ε, στην περιφέρεια της Ανατολικής Αφρικής. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του έτους, σε λίγους μήνες ελπίζουμε, να λανσάρουμε ε, την υπηρετική ζώνη ελευθερών συναλλαγών στην Αφρική, πράγμα που θα οδηγήσει σε δυνατότητα μετακίνησης εργαζομένων από μία χώρα, ακόμα και μία περιφέρεια της Αφρικής προς μία άλλη. Αυτό θα βοηθήσει τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης εντός Αφρικής και θα μειώσει και τον αριθμό εκείνων που ε, προσδοκούν να μεταναστεύσουν ε, περνώντας τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτό το πρόγραμμα ε, έχει συζητηθεί με συναδέλφους στις Βρυξέλλες και προσπαθούμε να βρούμε υποστήριξη διαφόρων αναπτυξιακών εταίρων για την εφαρμογή. Υπάρχει ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής, Παναφρικανικό μάλιστα. Συμπεραίνω. Στην εταιρική σχέση Ευρώπης-Αφρικής για τη μετανάστευση θα πρέπει να υπάρχει πιο έντονη συμμετοχή από πλευράς κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο παρελθόν υπήρχε ένας διάλογος αντίστοιχος, αλλά ήταν μάλλον μονόλογος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί συμμετέχουν πολλά κράτη-μέλη δικά μας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετέχει θα πρέπει να βελτιωθεί το καθεστώς θεώρησης διαβατηρίων για να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία στη διαχείριση, ανταλλαγή πληροφοριών, πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, του τράφικινγκ και προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταναστών προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων. Κατά πολέμηση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να οδηγεί σε μείωση της φτώχειας, ανάπτυξη και την ατζέντα μετά το 2015. Τελευταίο μου σχόλιο είναι αυτό που αφορά τις υποθέσεις τις εικασίας σε διάφορα έντυπα μέσα, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες την επεξεργασία και την ε, αντιμετώπιση των ε, ε, μεταναστών σε ορισμένες χώρες της Euromed. Τώρα, αν αυτό θα γίνει ή όχι στο εγγύς μέλλον, ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να, προσέχουμε στο μέλλον, αλλά από την αφρικανική άποψη αυτή η προσέγγιση που ακολουθεί όσα έχει προσπαθήσει να κάνει η Αυστραλία με την Παππούα Νέα Γουινέα, μπορεί όντως να δούμε να υποφέρουν από αυτή την κατάσταση τα δικαιώματα των μεταναστών σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη, για τις ενδιαφέρουσες σκέψεις σας. Επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Σπασία Παπαδοπούλου, που θα σχολιάσει τα αποτελέσματα του project για τους πρόσφυγες και τους εξόριστους. Κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και Εξορίστων είναι ένα δίκτυο 25 ΜΚΟ σε ολόκληρη την Ευρώπη που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των προσφύγων και των ετών των άσυλο. Πιστεύω πως ε, καταρχήν θα πρέπει να έχουμε τα εξής υπόψη μας όταν μιλάμε για πρόσφυγες, μετανάστευση και αναπτυξιακή βοήθεια. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο αριθμός των προσφύγων, ε, ε, ετών των άσυλο και εκτοπισμένων έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια. Είναι ένας τεράστιος αριθμός και η πλειοψηφία του δεν είναι στην Ευρώπη, ποτέ δεν θα έρθουν και ίσως και να μην θέλουν να είναι στην Ευρώπη. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι ο χρόνος που περνούν οι πρόσφυγες στην εξορία είναι περίπου 20 χρόνια και αυτό, μιλάμε, ε, και αυτό ονομάζεται παρατεταμένη κατάσταση πρόσφυγα. Δηλαδή είναι, πλέον δεν είναι θέμα ανθρωπιστικό, αλλά είναι θέμα ανάπτυξης και στήριξης μακροπρόθεσμων λύσεων. Θα ξεκινήσω με το γιατί χρειάζεται να στηρίξουμε τρίτες χώρες, ε, χώρες εταίρους ε, στο να αντιμετωπίσουν το θέμα των εσωτερικά εκτοπισμένων των προσφύγων. Καταρχήν, επειδή όλες οι χώρες, είτε είναι στην Ένωση είτε όχι, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις διεθνούς προστασία εφόσον έχουν υπογράψει διάφορες συμβάσεις ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο κόσμος θα πρέπει να μπορεί να προστατευτεί όπου βρίσκεται. Δεύτερον λόγο της αλληλεγγύης. Δηλαδή, δεν θέλει η Ευρώπη να μεταφέρει το πρόβλημα σε εκείνους ή να τους αφήσει να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους για να φιλοξενήσουν δηλαδή πρόσφυγες, αλλά γιατί όντως είναι σοβαρές οι προκλήσεις και πρέπει να στηριχθούν. Αλλά για να είμαστε αξιόπιστοι γι' αυτό θα πρέπει επίσης από την ευρωπαϊκή πλευρά να προσφέρουμε τη δυνατότητα να έρθουν εδώ με πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι, αν θέλουμε όντως αυτή η συνεργασία να είναι αξιόπιστη τρίτον, διότι ο εκτοπισμός είναι αναπτυξιακό ζήτημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τρόφιμα και κουβέρτες. Έχει να κάνει με την εξέβρεση λύσεων που θα βοηθήσουν τον κόσμο να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή από εδώ και στο εξή, ακόμα και αν είναι σε διαφορετικό μέρος από αυτό στο οποίο γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν. Καλωσορίζουμε τα πορίσματα του Δεκεμβρίου 2014 του Συμβουλίου, όπου ανέφεραν ότι οι ε, μεταναστευτικές ροές που προκύπτουν λόγω συγκρούσεων ε, και οι προκλήσεις που προκύπτουν από τους, πρόσφυγες, από τους πρόσφυγες και τους ιστορικά εκτοπισμένους αλλά και τους ετούντες άσυλο είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και είναι πολύ θετικό βρίσκουμε που αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Γίνεται επίσης λόγος για την ανάγκη εφαρμογής του Διεθνούς Πλαισίου Προστασίας. Εμεί μαζί με διάφορε ε, ε, ε, ΜΚΟ εταίρου έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα για την καλύτερη σύνδεση όλων αυτών των θεμάτων και ορισμένες συστάσεις για την αναπτυξιακή βοήθεια και θα ήθελα αυτά να τα μοιραστώ μαζί σας. Καταρχήν χρειάζεται συντονισμένη και, συντον, ε, συντονισμένη και συνεπής προσέγγιση. Δεν πρόκειται για το ε, διάφορες πολιτικές. Θέλουμε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη ε, καθολική προσέγγιση, ίσως να είναι πολύ κοινή λέξη τώρα τελευταία, αυτή η, κοινή, ολιστική, η ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πάντως αυτό θα πρέπει να γίνει για την αναπτυξιακή βοήθεια, την ανάπτυξη, αλλά και την εφαρμογή της ατζέντα ε, για την ε, ανοχή. Θα πρέπει να υπάρχει εταιρική σχέση και συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις, τοπικές αρχές. Η τοπική διάσταση είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί οι περισσότεροι πρόσφυγες ότι σήμερα ημέρα ζουν σε αστικές περιοχές. Δεν είναι σε στρατόπεδα, αλλά σε αστικές περιοχές. Επίσης θα πρέπει να δούμε τους πρόσφυγες ως οικονομικούς παράγοντες. Δεν είναι απλώς αποδέκτες βοήθειας. Συμβάλλουν στις τοπικές οικονομίες Ζουν, εργάζονται, ευημερούν, σπαταλούν, έχουν ε, ωφέλιμο αντίκτυπο στις ε, κοινωνίες στις οποίες ζουν. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία από αυτού και χρειάζεται να γίνει περισσότερη έρευνα ώστε αυτό να φανεί και να υποστηριχθεί. Επίσης πρέπει να στηρίξουμε τις ικανότητες των χωρών εταίρων να αντιμετωπίσουν τις τοπικές προκλήσεις δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για ε, ένταξη ε, και εδώ γι' αυτό χρειαζόμαστε στοχευμένες ε, παρεμβάσεις αλλά και προσχεδιασμό στις, στα πρώιμα στάδια μιας χρήσης. Τα δικαιώματα και οι ανάγκες των προσφύγων και των εκτοπισμένων χρειάζεται να ενταχθούν σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα και όχι μόνο ως στοχευμένη στήριξη για αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών. Τώρα όσον αφορά στοχευμένε παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στο νέο πλαίσιο, δημοσιονομικό πλαίσιο, το Ταμείο ε, Ασύλου ε, περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα για την προστασία των προσφύγων και για τη δημιουργία δυνατοτήτων στις τρίτες χώρες Επίσης το παγκόσμιο πρόγραμμα υπό το GCI έχει συμπεριλάβει ρητά τους πρόσφυγες οριζόντια ως ευάλωτες ομάδες σε διάφορα είδη ε, τομέων, δηλαδή κοινωνική προστασία, προστασία των παιδιών, Ίσως να πω δύο λόγια για τα προγράμματα περιφερειακής προστασίας ως στοχευμένη μορφή παρέμβασης, γιατί υπάρχει μια πρόθεση και ήδη έχει αναφερθεί στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, αλλά αναφέρθηκε και από τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και θα βρίσκεται στην ατζέντα για τη μετανάστευση, αλλά θα πρέπει ίσως να αναπτυχθεί περισσότερο. Και υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα, δηλαδή το πρόγραμμα ε, περιφερειακής προστασίας στη Μέση Ανατολή και έχουμε κάνει σχετική έρευνα όσον αφορά τα περιφερειακά προγράμματα προστασίας από το 2005 μέχρι τώρα ε, και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι μέχρι στιγμής ε, ήταν κατακαιρματισμένα και μερικά αυτά τα προγράμματα είχαν κάποιο αντίκτυπο σε κάποιες περιπτώσεις υποστηρίχθηκαν ε, υποστηρίχθηκε η προστασία, αλλά σε άλλες περιπτώσεις απλά στην ουσία σήμαινε κάποια βασική επιπλέον μάλλον χρηματοδότηση ώστε το, η υπατερμοσία για τους πρόσφυγες να συμπληρώσει κάποιες βασικές ανάγκες. και αυτό γιατί ήταν μικρά τα προγράμματα, περιορισμένη χρηματοδότηση. Έπειτα υπερβολικά πολλοί στόχοι σε κάθε μικρό προγραμματάκι που δεν μπορούν να υλοποιηθούν έλλειψη συνοχής με άλλες παρεμβάσεις στην ίδια χώρα, έλλειψη συντονισμού με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που γίνονται στην ίδια χώρα και που θα μπορούσαν να στηρίξουν γενικά τις ανάγκες των προσφύγων και των ετούντων άσυλο και το πιο σημαντικό είναι η έλλειψη της εμπλοκής των χωρών εταίρων ώστε να αντιμετωπίσουν και να στηρίξουν τις ανάγκες των εκτοπισμένων και των προσφύγων. Γι' αυτό και χρειάζεται και πολιτικός διάλογος. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, άρα αν είναι μέρος του πολιτικού διαλόγου με τις χώρες εταίρες. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο για να μιλήσω για την τον παρατεταμένο εκτοπισμό. Είπα ότι ορισμένοι άνθρωποι μεγαλώνουν σε στατόπεδα προσφύγων, ζουν εκεί για 20 χρόνια και ακόμα εξεκολουθούμε να το θεωρούμε αυτό ως ανθρωπιστικό ε, ε, θέμα, ενώ είναι αναπτυξιακό. Συστηματικά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ο παρατετημένος εκτοπισμός στις ε, αναπτυξιακές στρατηγικές και να αναζητήσουμε τρόπους με τους οποίους ο κόσμος αυτός θα μπορούσε να προχωρήσει, να έχει πρόσβαση στην παιδεία, στην κατάρτιση, στην αυτάρκεια εκεί όπου βρίσκεται ή στις γειτονικές χώρες και το πλαίσιο για κοινοτικότητα ε, που ανεφέρθη από τον κύριο Πρέσβη δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες για κινητικότητα που μπορεί να στηρίξει και την αυτάρκεια και τις πιο μόνιμες λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπαδοπούλου και τώρα να ακούσουμε τον Γενικό Διευθυντή του Solidar, τον κύριο Ρόιτερ. Θα είναι σημαντικό να ακούσουμε τι γίνεται στο ιστορικό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Solidar για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα πρέπει να σας πω ότι μου προκαλεί θετική εκπλήξη η σημερινή ημέρα. Γιατί από το μετρό που ήρθα μέχρι εδώ δεν είχε κόσμο και έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ στην αίθουσα για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τον ενδιαφέρον σας. Και όπως ξέρετε, οι, οι Αμερικάνοι πολιτικοί μιλάνε για κατάσταση και προσέγγιση win-win, εποφελούσα ε, ωφέλους. Αλλά συχνά όταν μιλάμε για την μετανάστευση δεν μας υποστηρίζει η πλειοψηφία. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το φετινό έτος γιατί θα γίνει η συζήτηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έτους για την ανάπτυξη. Το θέμα είναι λοιπόν ε, τα όμορφα λόγια για την ε, συνοχή, για την ανάπτυξη και τις σχετικές πολιτικές ε, είναι τόσο θεωρητικά όσο και η ολιστική προσέγγιση, η συνολική προσέγγιση. Παντού ε, ξεφυτρώνει αυτή η έκφραση. Τι σημαίνει όμως αυτό όταν μιλάμε για μετανάστευση, ποιοι είναι οι... Ποιες είναι οι αιτίε που προσελκύουν και σπρώχνουν τους ανθρώπους εκτός, από τις, εκτός των χωρών τους. Οι χώρες που διώχνουν τους ανθρώπους είναι η κοινωνική και οικονομική κατάσταση, ο κίνδυνος στην ε, επιβίωσή τους. Όπως ε, η κυρία Κέλλερ ε, στις 3 Οκτωβρίου είδαμε την κατάσταση στην Λαπεντούζα και δεν επισκεφτήκαμε ένα όμορφο νησί στην Μεσόγειο, αλλά προσπαθήσαμε να σκεφτούμε για ένα λεπτό τι μπορεί να σπρώχνει τον κόσμο να μπει σε αυτά τα βαρκάκια. Θα πέρατε ένα τέτοιο μπουκάλι νερό για να πάτε να περάσετε στη Μεσόγειο σε ένα βαρκάκι. Τι σπρώχνει λοιπόν τον κόσμο να το κάνει αυτό. Ο φόβος για τη ζωή τους θέλουν να έχουν μια αξιοπρεπή δουλειά, μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτό αποτελεί το βασικό ζήτημα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να, όχι μόνο να μιλάμε για το Frontex, για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, αλλά αν δεν φροντίσουμε τον κόσμο να έχει μια αξιοπρεπή ζωή, ούτε το τείχος του Βερολίνου δεν απέτρεψε τον κόσμο από το να κινείται από την Ανατολή προς τη Δύση. Λοιπόν, πώς μπορούμε να βρούμε ανθρωπιστικές λύσεις, από την άλλη και οικονομικές λύσεις και να βρούμε κυρίως κοινωνικές λύσεις. Αυτό που είπε ο κύριος Αμβρόζη, καταρχάς, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη τις πραγματικότητες. Δεν μιλάμε για τον παράγοντα του φόβου. Μιλάμε για τόσο μεγάλα, τόσα πολλά εκατομμύρια μεταναστών. Ξέρετε ότι λίγοι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και μιλάμε για 32 εκατομμύρια. Βλέπετε από το 233 εκατομμύρια των μεταναστών πόσο μικρό ποσοστό είναι τα 32 εκατομμύρια. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στο Μεξικό. Ε, είναι κόσμος ε, νέοι κυρίως οι οποίοι ανεβαίνουν στα τρένα, πάνω στα τρένα δηλαδή και προσπαθούν από την, κεντρική, από την ε, Νότια Αμερική να περάσουν την Κεντρική Αμερική να πάνε στο Μεξικό για να φτάσουν στη ΣΥΠΑ. Ούτε καν ένα μπουκάλι νερό δεν έχουν. Εδώ και τέσσερις δεκαετίες λοιπόν το θέμα της μετανάστευσης μας απασχολεί όλο. Βγαίνουμε και λέμε ότι θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, έχουμε ανάγκη το ένα, έχουμε ανάγκη το άλλο. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για συνοχή στις πολιτικές μας, θα πρέπει να αποδεχτούμε πιο αποτελεσματικές ότι οι πιο αποτελεσματικές πολιτικές ανάπτυξης δεν θα σταματήσουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές, γιατί μεταξύ της επένδυσης σήμερα και του αντίκτυπου θα περάσουν πολλά χρόνια. Και από την άλλη πλευρά της Μεσογείου, αν δούμε τι γίνεται στις χώρες αυτές, πού είναι η οικονομική ανάπτυξη, πού είναι η δυνατότητα να, που θα είχε ενδεχομένω ο κόσμος να μείνει στις χώρες τους και να δουλέψει. Και αυτό με φέρνει στο επόμενο ζήτημα. Μπορούμε να συζητάμε ανθρωπιστικές λύσεις, αλλά θα πρέπει να συζητάμε και οικονομικές λύσεις. Οι οικονομικές ε, λύσεις έχουν να κάνουν με μια σωστή ατζέντα για την απασχόληση. Το ίμιση και άνω των μεταναστών φεύγουν από τις χώρες τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν, γιατί δεν έχουν μία αξιοπρεπή δουλειά. Πρέπει να φροντίσουν λοιπόν να έχουν ένα κάποιο εισόδαμα, να έχουν ε, τρόφιμα, να μπορούν να τρέψουν την οικογένειά τους. Αυτός ο σύνδεσμος λοιπόν ε, με την ε, πολιτική για την απασχόληση του ΠΟΕ είναι πολύ σημαντικός και αν μιλάμε για τις ευκαιρίες που έχουμε στην τρέχουσα χρονική συγκυρία είναι δύο. Καταρχάς, να μιλήσουμε για την επένδυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσιάζει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης και θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε την επένδυση σε ε, συστήματα κοινωνικής προστασίας γιατί αυτό θα προστατεύσει τον κόσμο. Η προστασία δεν αποτελεί προσβολή, αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Γι' αυτό λοιπόν η επένδυση σε βασικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας είναι πολύ σημαντικό στο ιστορικό της Ευρώπης. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη χρονική συγκυρία, φέτος το καλοκαίρι, είναι το συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας στη Γενέβη το καλοκαίρι. Πώς μπορούμε λοιπόν να συμβάλλουμε στη δημιουργία μια σωστή οικονομικής και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ε, στις χώρες ε, τις γειτονικές, στην άλλη πλευρά της Μεσογείου. Είναι σημαντικό να βρούμε λύσεις, να σκεφτούμε το πώς μπορούμε να επενδύσουμε για να δημιουργήσουμε σωστές ε, και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίες. Στην όλη αυτή τη συζήτηση ακούμε διάφορα για την προσέγγιση βάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ απαραίτητο γιατί ο πολιτισμός μας διαφέρει από τους άλλους στην ρού της ιστορίας γιατί υπάρχει ακριβώς αυτή η αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κρατός δικαίου και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να ερμηνευτεί με τρόπο που να περιλαμβάνει και τους μετανάστες, είτε είναι νόμιμοι είτε είναι χωρίς χαρτιά. να υπάρχει αυτή η προσέγγιση βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοιτώντα τι γίνεται στι χώρε προέλευση κάποιων μεταναστών και προσφύγων ιδιαίτερω, βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθηθεί και αυτή η ιδέα στην κοινή γνώμη ότι έχουν αναπαλωτρίωτα δικαιώματα. Αυτό είναι απαραίτητο. Η πρόεδρος Λίντα Μακέβαν είπε στην αρχή κατά πόσον έχουμε λύσεις. Αν είχαμε λύσεις δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τι χρειάζεται. Χρειάζεται καταρχάς τόλμη και αποφασιστικότητα. Πρέπει να, βγει, να βγούμε και να προασπίσουμε την ιδέα αυτή ότι χρειαζόμαστε αυτές τις πολιτικές και πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Και με το, την τόλμη και το θάρρος εννοώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε και οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι πολύ δημοφιλείς. Αν δεν θέλουμε να συνεχιστεί το τράφικινγκ, να μείνει με την αβεβαιότητα ο κόσμος και με τον κίνδυνο που διατρέχουν, θα πρέπει να σκεφτούμε πρακτικές λύσεις οι οποίες δεν θα είναι δημοφιλείς. Ο, η λύση ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου θα πρέπει να τύχει διαπραγματεύσεις, γιατί θα συνεχίσουν να έρχονται Άρα, καλό θα ήταν να μην μιλάμε μόνο για μια κουλτούρα υποδοχής, αλλά να αποδεχτούμε ότι ο κόσμος αυτός χρειάζεται κάποιες συνθήκες για να μπορεί να έρχεται εδώ. Με τον ανθρωπιστικό διάδραμο έχουμε και ένα πολιτικό εργαλείο, όχι πολιτικό όπλο, αλλά πολιτικό εργαλείο για να διαπραγματευόμαστε με τα κράτη-μέλη, για να λέμε ότι κοιτάξτε αυτό δεν είναι ένα θέμα που πλήττει μόνο την Ευρώπη, την, Ισπα... την Ιταλία, την Ισπανία, αλλά όλη την Ευρώπη και τα 28 κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό λοιπόν να διαπραγματευτούμε και να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα και να πούμε ότι έτσι θα προχωρήσουμε. Νομίζω ότι δεν έχω και άλλο χρόνο, αλλά ας πούμε μια τελευταία κουβέντα για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Αν δεν θέλουμε να έχουμε μόνο τα όμορφα εγγένεια στη, όπως είχαμε στη Ρήγα με φανταστικές ομιλίες θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτό το Ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης, πώς μπορούμε να, προκαλέσουμε, να αποτρέψουμε τη σύγχυση με τις εμπορικές πολιτικές, πώς μπορούμε να δώσουμε νόημα σε κάτι που έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Επενδύσεις ευφυείς που θα επιτρέψουν στον κόσμο να μείνει εκεί που είναι και να έχει μια αξιοπρεπή ζωή. Και επίσης ας συνδέσουμε και τον ε, Επιτροπό Τίμερμανς, ο οποίος ε, έχει απευθύνει τέτοιες ε, ωραίες ομιλίες και έχει απευθυνθεί και στον κύριο Στόιμπερ τη Βαβαρία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως θα μπορούσε να θέσει και το θέμα τη ανάπτυξη και τη μετανάστευση βάσει τη προσέγγισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό δεν αποτελεί μόνο ένα όνειρο, μια όμορφη ομιλία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αλλά όπω σα είπα αυτό χρειάζεται και προαπαιτεί τόλμη αποφασιστικότητα. Και για να σας ε, βάλω και στη σωστή διάθεση. Κοιτάξτε εν ώψη του Πάσχα στο iPhone σας. Ε, σας συστήνω δύο τραγούδια, του Μανούτσα ο Κλαντεστίνο, το ένα και το άλλο για ηλικιωμένους του 69, Led Zeppelin, The Immigrants. Led Zeppelin. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε αυτή την τόλμη για να δράσουμε πραγματικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας παρουσιάσατε αυτά τα στοιχεία, να τα σκεφτούμε, κάποιες ενδεχόμενες λύσεις μέσα σε αυτές. Αν και κάποιες από αυτές τις λύσεις είναι πολιτικώς δύσκολες. Ίσως θα ήθελαν οι συνάδελφοι να αυτοσυστήνονται όταν παίρνουν το λόγο, γιατί δεν είμαστε μέλη της ίδιας επιτροπής όλοι. Αν θα θέλετε λοιπόν να κάνετε μια εισαγωγή για να παρουσιάσετε το θέμα σας και να συστηθείτε. Αν θα θέλετε να σηκώσετε τα χέρια σας για να δούμε πόσους ομιλητές έχουμε και να δούμε και πόσο χρόνο λοιπόν θα έχει ο καθένας. Γιατί έχουμε 50 λεπτά στη διάθεσή μας. 2 έως 3 λεπτά. 2 λεπτά, 2 λεπτά ο καθένας, μου λέει η συμπρόεδρος. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ και μετά η κυρία Βίμπεργκ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χουάν Λόπεθ Αγγιλάρ, είχα τη χαρά να συναντηθώ με κάποιους από τους προσκεκλημένους και ομιλητές μας σήμερα το πρωί. Πολύ καλή η ανταλλαγή απόψεων και τη χειροκροτώ. Είμαστε όλοι στεναρά πεπισμένοι, είτε είμαστε μέλη της Επιτροπής Ελευθεριών, είτε της Επιτροπής Ανάπτυξης, ότι το άσυλο συνδέεται με την ανάπτυξη και τούντες άσυλο δεν είναι απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τράφικε γίνεται. Έχει να κάνει όμως και με τη μετανάστευση αυτό το θέμα, γιατί πολλοί από τους λεγόμενους παράτυπους μετανάστες θέλουν μια ευκαιρία στη ζωή τους. Ξεφεύγουν από την απομόνωση, από αφόρητες καταστάσεις, από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι μεγάλη πρόκληση η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι παγκόσμιο πρωταγωνιστής, player, παίκτη είναι της μόδας να λέμε, και όχι μόνο payer, πλήρωτης. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αμπρόση, με τον οποίο έχω συναντηθεί όπως σας είπα και στο γραφείο μου ως μέλος επιτροπή Επιτροπής Ελευθεριών για θέματα μετανάστευσης. Ε, εκπροσωπεί το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση για την Ευρώπη. Ακούσαμε για μια πρόταση και βλέπουμε και από τα διεθνή δημοσιεύματα στον τύπο που λέγει ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι σκέφτονται να αναθέσουν ε, σε κάποιους εξωτερικούς της επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο και ψάχνουν προτάσεις να δημιουργηθεί ένας τρόπος, ένα σύστημα πραγματικής αποτροπής για να έρχονται να έρχονται λιγότεροι μετανάστες στις ευρωπαϊκές ακτές. Υποθέτω ότι έχει συζητηθεί στο περιθώριο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και ορισμένοι υπουργοί έδωσαν συνέχεια στην πρόταση αυτή και την ε, συζητούν σε διάφορα Υπουργεία Εσωτερικών ε, ακόμα και καταβλισμοί προσφύγων να ε, μετακατασταθούν σε χώρες όπως η Τινησία και η Αίγυπτος. Τι λέει το Γραφείο Μετανάστευσης για αυτά τα θέματα, για τη συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό εγγράφεται ή όχι ε, στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ευθυγραμμίζεται με όλες αυτές τις αρχές και τις μη επαναπροώθησης. Ε, ακόμα και με τις συστάσεις που έχουν γίνει από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Η κυρία Βίμπερκ και μετά η κυρία Βίξου. Ε, ε, σας ευχαριστώ. Η ανάπτυξη και η μετανάστευση είναι ενδιαφέρον, αποτελούν ενδιαφέρον συνδυασμό. Πάντα είχαμε μετανάστευση. Το θέμα είναι τι ποσότητα μετανάστευσης, τι όγκο μετανάστευσης χρειαζόμαστε. Να σας μιλήσω για τη δική μου χώρα. Είδαμε ότι χρειαζόμαστε μεταναστευτικές ροές για να αντισταθμίσουμε τις ε, ανάγκες για τα συνταξιωτικά συστήματα. Αλλά στο παρελθόν έχουμε μεγάλα ε, προβλήματα, είχαμε μεγάλα προβλήματα και σε ό,τι αφορά την ανεργία. Η μαζική λοιπόν ανεργία, η μαζική σε μετανάστευση οδήγησε σε ανεργία. Και τώρα λοιπόν ε, έχουμε συγκεκριμένες ποσοστώσεις ε, για τη μετανάστευση. Έχουμε περιοχές όπου έχουμε πολλές μετανάστες στη Σουηδία, όπου υπάρχουν βία περιστατικά και αυτοκίνητα και σχολεία. Μεγάλες μεταναστευτικές ροές εκεί, υψηλή ανεργία και όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Παράνομη μετανάστευση, λάθρο μετανάστευση, μεγάλα ποσοστά στη Σουηδία. Υπάρχουν βέβαια τα κοινωνικά δικαιώματα και στις περιπτώσεις αυτές, ακόμα και αν δεν έχει λάβει κανείς ε, άδεια να παραμείνει. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κατανάλωση γιατί αγοράζει ο κόσμος αυτός, αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ε, λάθος μηνύματα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι επιρροές στην ε, Σουηδία. Ευχαριστώ, κυρία Στυρ. Κύριε Βίξτρομ και μετά κύριο Στυρ. Στήρ. Ευχαριστώ. Πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας λέτε και ε, εκτενή. Δεν ακούμε πάντα στο Κοινοβούλιο μιλητές ε, με τόσο ενδιαφέροντα πράγματα να μας πούν για το τι συμβαίνει. Ανεξαρτήτως του τρόπου διάσωσης που θα επιλέξουμε, όπως είπε ο κύριος Ρόιτερ, θα έρχεται ο κόσμος με ένα μπουκαλάκι νερό και τίποτα άλλο. Ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι να ε, σπάσουμε αυτή την πίσνα των διακινητών, να μην είναι κερδοφόρο, ή να μην ε, ε, σκυλοπνίγονται οι άνθρωποι στη Μεσόγειο σε αυτά τα σκάφη που κινδυνεύει να γίνει τεράστιο νεκροταφείο η Μεσόγειος. Κάθε χρόνο χιλιάδες πνίγονται προσπαθώντας να φτάσουμε ναι, στις αρχές μας, τακτές μας. Τι σημαίνει να τους σπάσουμε την πίσνα, να σπάσει το μονοπόλιο τους και να το δούμε με έναν τρόπο αξιοπρεπή. Θα ήθελα να το συνδέσω και με το θέμα ασφαλείας. Σήμερα όλοι εδώ μέσα και στην Ευρώπη συζητούν για θέματα ασφαλείας. Εάν επιτρέπουμε στον κόσμο να έρθει με τρόπο συντεταγμένο, προστατευμένο, ασφαλή σε κάποια κράτη ή σε ένα κράτος και να υποβάλει αίτηση ασύλου, θα ξέρουμε ακριβώς ποιος έρχεται, από πού έρχεται και υπό ποιες συνθήκες. Και αυτό συνδέεται με το θέμα ασφαλείας που απασχολεί τους πάντες και το συζητούν όλοι σήμερα. Εμείς θα πρέπει όμως να προσφέρουμε μία εναλλακτική λύση. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Ένας τρόπος είναι να συμμετέχουν περισσότερα κράτη-μέλη στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΥΠΑ της Αρμοσίας για τους πρόσφυγες και να ξανακοιτάμε τις αιτήσει ασύλου, ας πούμε, σε προσωρινά γραφεία στους καταβλισμούς προσφύγων. Έξι κράτη-μέλη σήμερα λαμβάνουν 80% των των άσυλο. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την αλληλεγγύη δια νόμου, αλλά χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη, όχι μόνο μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών. Ερωτώ, θα υποστηρίζατε ένα σύστημα ποσοστώσεων, η ερώτηση απευθύνεται προς όλους, για να αυξηθεί ε, ο επιμερισμός της ευθύνης μεταξύ κρατών μελών. Κύριε Πρέσβη, εσείς πώς βλέπετε τη συνεργασία με τις λεγόμενες ασφαλείς τρίτης χώρες. Και τι γίνεται με ε, την επεξεργασία αιτήσεων ασύλου σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Steer followed by Madam Hautala. Thank you, Madam Chair. Thank you to all the speakers. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Θα προχωρήσω σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα και μια ερώτηση. Η χώρα μου ε, η χώρα που γνωρίζω καλύτερα επειδή γεννήθηκα εκεί είναι η Αργεντινή και είναι μια χώρα στην οποία, ε, της στο Σύνταγμα ε, υπάρχει κάτι το, που είναι φτιαγμένο για να προσελκύσει μετανάστες κυρίως από την Ευρώπη και αυτό έγινε με, όταν η κατάσταση ήταν ευημερής όταν άρχισε να ανθεί η διαφθορά δυστυχώς στη χώρα και η χώρα άρχισε να προχωρά πολύ πιο αργά και τώρα είναι μια χώρα ε, που, ε, από την οποία φεύγει, ο κόσμος. Με βάση αυτό το παράδειγμα λοιπόν, η ερώτησή μου είναι σε όλους τους ομιλητές, όταν θα έχουν ε, το λόγο για να απαντήσουν, είναι αν μπορούν να συμπεριλάβουν την σχέση ανάμεσα στην ε, στους θεσμούς και την δημιουργία αυτών, αυτής της κατάστασης. Εμείς έχουμε, ας πούμε, ε, ε, αυτό τον προβληματισμό. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους θεσμούς μας ώστε να βελτιώσουμε και την αναπτυξιακή μας βοήθεια κατά συνέπεια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάουταλ, ε, ήταν πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε για το θετικό αντίκτυπο των ε, του, του, του ενδοαφρικανικού και περιφερειακού εμπορίου καθώς και την ε, ελεύθερο εμπόριο. Ιδιαίτερα πιστεύω ότι οι, οι συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας μπορεί να δημιουργήσουν προκλήσεις και δυσκολίες, ενώ αυτού του είδους εταιρικέ σχέσεις και οι περιφερειακοί σχέσεις είναι ε, πολύ και ε, είναι πολύ καλό το παράδειγμα της, Ένωσης ε, Κρατών της Ανατολικής Αφρικής Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, θα αναπτυχθεί περισσότερο αυτή η σύνδεση. Το ερώτημα μου είναι, σε σχέση με αυτό το New Deal του 2011, ε, μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει πώς αυτή η εταιρική σχέση με τα ευάλωτα κράτη, ώστε να βοηθήσουμε την οικοδόμηση κρατών και, και ειρήνης, μπορεί να βοηθήσουν για στις μεταναστευτικές ροές που συχνά προκαλούνται λόγω ε, βίας, εχθρικής και τοπικής κοινωνίας κυρία Κέλλερ και μετά η κυρία Σράιν. Έχω κάποια σχόλια και κάποιες ερωτήσεις. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι συχνά όταν μιλάμε για ανάπτυξη και μετανάστευση, ε, αυτό που κοιτούμε είναι οι χώρες ε, αποδέκτες, ε, οι χώρες προέλευσης. Και εγώ είμαι από μια περιοχή που ήταν μεταναστευτική περιοχή. ο κόσμος ακολουθούσε την κοινή λογική όταν πήγαινε κάπου, γιατί δεν μπορεί να περιμένεις ο κόσμος να περιμένει 20-30 χρόνια μέχρι να αναπτυχθεί η περιφέρειά τους. Και έπειτα είναι στο προσωπικό συμφέρον να κάνει κανείς αυτή την κίνηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ατομική ανάπτυξη. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο για τις κλιματική, την κλιματική μετανάστευση. Και αυτός είναι ένας βασικός ε, παράγοντας ε, νότου, για τη μετανάστευση νότου-νότου. Το κλίμα ε, συχνά δεν καταλήγουν εδώ, καταλήγουν αλλού. Πηγαίνουν στην επόμενη περιφέρεια, την επόμενη χώρα και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί και οι χώρες όπου πηγαίνουν είναι χώρες υπό ανάπτυξη. Το θέμα είναι λοιπόν πώς στηρίζουμε αυτές τις χώρες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα μέχρι να αναπτυχθεί κάθε περιοχή, αλλά και σε εκεί που εξαφανίζονται ολόκληρα νησιά και τα προβλήματα που προκύπτουν από εκεί. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει, αλλά σε άλλες όχι. το θέμα των εξωτερικών ε, στρατοπέδων προσφύγων ε, και της διάσωσης και εγώ είμαι κατά του, αυτού του συστήματος αλλά βέβαια αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν υπάρχουν χώρες που θέλουν να φιλοξενήσουν αυτά τα στρατόπεδα προσφύγων και να πούνε ναι εμείς παίρνουμε χρήματα από την Ένωση και συμβάλλουμε στο θέμα αυτής της εξωτερήκησης ε, τι, τι λέτε εσείς στην Αφρικανική Ένωση υπάρχουν χώρες που θέλουν να παίξουν αυτόν τον ρόλο, που επαναλαμβάνω εγώ δεν είμαι καθόλου σύμφωνη με αυτόν. Τώρα, το θέμα των ποσοστώσεων θα έλυνε ίσως το μισό το πρόβλημα που έχουμε, το πρόβλημα της αλληλεγγύης, αλλά μετά ξεχνάμε το θέμα του μεμονωμένου μετανάστη που μπορεί να έχει διαφορετικό ενδιαφέρον για να πάει κάπου αλλού. Να, συγγνώμη, πρέπει να κλείσετε τώρα, λέει η Πρόεδρος. η κυρία Σφάι. Σλάι. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ που θυμήσατε και τη Λαμεντούζα, γιατί ήμουν και εγώ εκεί τον περασμένο Οκτώβριο. Είναι απίστευτο που πρώτα φτιάξαμε ένα κοινό ευρωπαϊκό νεκροταφείο αντί να φτιάξουμε ένα κοινό σύστημα ευρωπαϊκό που είναι απαραίτητο για να βρούμε λύσεις. Και επίσης θυμήσατε ότι, και σας ευχαριστώ ότι δεν είναι πρόβλημα της Ιταλίας, της Μάλτας ή της Ελλάδας, είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό. Και γι' αυτό πρέπει να βρούμε λύσεις. Συχνά στην Ιταλία μας ρωτάνε μα πού είναι η Ευρώπη μπροστά στην Λαμπεντούζα. Αν δούμε τα στοιχεία για τα αιτήματα ασύλου, μόνο έξι χώρες ε, ε ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ε, οι υπόλοιπε κυβερνήσει που είναι. Αυτή είναι η αλληλεγγύη για την οποία μιλά το άρθρο 80 της συνθήκης. Συμφωνώ ότι πρέπει να βρούμε μια βραχυπρόθεσμη λύση αλλά και μια μακροπρόθεσμη λύση. Η βραχυπρόθεσμη δεν μπορεί παρά να είναι το να κάνουμε πιο σύντομα τις παρεμβάσεις να κάνουμε μελέτες για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, για να δημιουργήσουμε δηλαδή νόμιμες οδούς και ασφαλείς οδούς για τους πρόσφυγες αλλά και για τους μετανάστες Επίσης θα πρέπει να καταπολεμηθούν οι ανισότητες. Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης και ευχαριστώ τον Αμπρόζη που το τόνισε αυτό, ότι είναι πολύ μεγάλη σύνδεση ανάμεσα στην μετανάστευση και τις ανισότητες. Επί τις πιο αποτελεσματικές αναπτυξιακές πολιτικές, να επιμείνουμε σε καλύτερη κινητοποίηση των εγχώριων πόρων, να μπορέσουμε δηλαδή να σταματήσουμε τις παράνομες ροές ε, ε, κεφαλαίου, το θέμα της φοροαποφυγής στις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι πραγματικά οι παράνομες ροές κεφαλαίου είναι πολύ πιο μεγάλες από ότι η ροή βοήθειας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι οι φιλόδοξες αυτές ε, λύσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, θα πρέπει κάπως να μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή. Ευχαριστώ η κυρία Χορμπρούκ και μετά η κυρία Λόριστην. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που δεν διεκπαιρέωσαν το θέμα αυτό μόνο από λειτουργική και γραφειοκρατική άποψη, γιατί πάντα κρύβεται μια ανθρώπινη ιστορία με μια ανθρώπινη διάσταση πίσω από τα θέματα αυτά. Και είναι καλό λοιπόν το οποίο το έχουμε, το έχουμε αυτό υπόψη. Θα ήθελα καταρχά να υποστηρίξω την ιδέα του ανθρωπιστικού διαδρόμου και εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο ω μέτρο, γιατί είναι καλό μέτρο να ε, καταπολεμήσουμε το τράφικινγκ και τους λαθρεμπόρους ανθρώπων. Και ναι, αλλά έχουμε και λίγο ποιοι άνθρωποι έρχονται πού έρχονται. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να το τονίσω εδώ. Κάτι άλλο να αναφέρω. Αναφέρεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αναφέρεται εκ νέου η πολιτική συνοχή και ο συντονισμός. Αναρωτιέμαι. Πού είναι η πολιτική συνοχή στην πράξη? Ένα μικρό παράδειγμα να δώσω. Κλείνουμε τα σύνορα στην Ευρώπη, αλλά οι μετανάστες που είναι εδώ και έχουν θέσεις απασχόλησης υποστηρίζουν τις οικογένειάς τους, τις πατρίδες τους και είναι ένα μεγάλο τμήμα του, των χρημάτων που περιλαμβάνονται στην ανθρωπιστική βοήθεια και την αυτοξιακή βοήθεια. Αυτά που δίνει ο κόσμος στην οικογένειά του, στην πατρίδα του αυτό που ενδεχομένως χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτήσει και τους λαθρεμπόρους ανθρώπων, τους διακινητές. Πρόκειται λοιπόν ε, για ανεπίσημες, άτυπες μορφές ε, ροών χρημάτων. Εδώ λοιπόν γιατί δεν έχουμε πολιτική συνοχή. Γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα τέτοιο παράδειγμα. Θα ήταν λοιπόν λογικό να δημιουργήσουμε επίσημες οδούς ε, για να δούμε τι ροές χρηματικές υπάρχουν και πόσο έντονη και μεγάλη είναι η υποστήριξη προς τις οικογένειές τους. Όταν μιλάμε λοιπόν για πολιτική συνοχή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ε, νομική θέση των μεταναστών στις χώρες μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόιστη και κυρία Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία έθεσε τη διάσταση της ε, συνολικής προσέγγισης και έθεσε το θέμα υπό ευρία έννοια, γιατί είπατε 20 χρόνια αναφέρατε. Αυτό τι σημαίνει ως μεσόωρο ότι η στιγμή που καταφτάνουν είναι μία στιγμή. Αλλά μετά ακολουθεί μία μακρά περίοδο. Και το θέμα λοιπόν που ανακύπτει είναι πώ αυτό ο κόσμο θα βρει τρόπο να ενταχθεί, να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή κοινωνία, στι τοπικέ κοινωνίε. Και εδώ πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε μία στιγμή. Για τη συνολική στρατηγική βλέπουμε εδώ ότι το επόμενο έτος τα κονδύλια για την ανάπτυξη θα είναι 203 εκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει ότι στα κονδύλια αυτά θα πρέπει να δούμε τι αφιερώνεται στην ενσωμάτωση στην παιδεία, όχι μόνο εκπαίδευση για επαγγελματικές ικανότητες. Θα πρέπει να σκεφτούμε πιο πολύ την ευρωπαϊκή προσέγγιση σε τέτοιου είδου ενσωμάτωση, εκπαίδευση, παιδεία, όχι μόνο την ώρα που φτάνει ο κόσμος αλλά και την φάση ένταξής του. Ο κόσμος που καταφθάνει μπορεί να προστατεύεται από τον νόμο. Αλλά αν δεν συνεργαστεί η τοπική κοινότητα, αν δεν αντιληφθεί η τοπική κοινότητα τα δικαιώματά του, θα υπάρχουν συγκρούσει. Μοιραία. Στο Παρίσι, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι οι νέοι που έχουν γεννηθεί, έχουν γαλοχηθεί στην Γαλλία, τελικά γίνουν δολοφόνοι. Αν δούμε το θέμα των Αλβαπών μαχητών, βλέπουμε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο παίρνει όλο και πιο μεγάλο διαστάση. Θέλουμε λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την παιδεία και τον αντίκτυπο της παιδεία. Θα πρέπει να υπάρχει διαπολιτισμική διάσταση, θα πρέπει να περιλαμβάνει πιο πολλέ ε, πολιτισμικέ ε, διαστάσεις. Πόσα άτομα εργάζονται στις οργανώσεις αυτές που ασχολούνται με τους πρόσφυγες μετανάστες ετούντες άσυλο. Πόσες θέσεις θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για τον κόσμο αυτό που εργάζεται με τα άτομα αυτά. Τους Ρωμά συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Επί δεκαετίες δεν βρίσκουμε λύση στο θέμα αυτό και πάλι αυτό έχει να κάνει με την ένταξη, με την παιδεία, την εκπαίδευση. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Αυτό τώρα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρχει και ευρωπαϊκή διάσταση στην ευθύνη αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Μάγια και Σαρχεντίνη στη συνέχεια. Μέγερ, πώς σας λένε, μπορείτε να μου πείτε. Πολύ ωραία, το είπατε Μάγερ και σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ερώτησή μου απευθύνεται στον κύριο Αμπρόζη. Σας άκουσα να ζητάτε αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μαζική λαθρομετανάστευση. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αυτή την έκκληση την απευθύνεται και στις χώρες της, της περιφέρειας από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες για να είναι καλύτερη η υποδοχή τους στην περιφέρειά τους αντί να έρχονται εδώ. Άκουσα και κάποιους ομιλητές να κάνουν λόγο για τις συνέπειες που έχουν για τις χώρες από τις οποίες ε, αποχωρούν. Έχετε σκεφτεί τι συνέπειε που έχουν για όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες για τις χώρε που καλούνται να του υποδεχθούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρχεντίνη και μετά ο κύριο Γκερέρο Σαλόν. Σα ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον στη συζήτηση για τη μετανάστευση στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι το πόσο Ευρωπαίοι το πρόβλημα της μετανάστευσης, γιατί κυρίως ως πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε, το κάνουμε outsourcing σε τρίτες χώρες, το αναθέτουμε εξωτερικά. Για παράδειγμα, να το θέσω αυτό ως παράδειγμα σε σχέση με αυτό που είπε ο πρεσβευτής της Αφρικανικής Ένωσης για τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη για το πώς μπορούμε να κρίνουμε το θέμα της μετανάστευσης εκτός των συνόρων μας και θα συμφωνήσω με την ε, συνάδελφο Σκάι ότι εγώ δεν συμφωνώ. Ένα άλλο παράδειγμα για το οποίο πήρατε εσείς την πρωτοβουλία και όπου οι ευρωπαϊκές χώρες ε, συμφωνούν και συνδράμουν είναι η διαδικασία του μου. Και πολύ λυπάμαι, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται τη στιγμή που τα ευρωπαϊκά κράτη ε, με την Ερυθρέα, το Σουδάν, την Αιθιοπία και άλλα αφρικανικά κράτη έχουν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι μεγάλοι προμηθευτές, αν θέλετε, αυτές οι χώρες ε, πολιτικών προσφύγων. Και λοιπόν τα ευρωπαϊκά κράτη ε, έχουν συμβάσεις και συμφωνίες με τις χώρες αυτές. Και θεωρώ ότι έτσι ουσιαστικά κάνουμε μια ευρωπαϊκή, από ευρωπαϊκή πλευρά μια εξωτερική ανάθεση του προβλήματο. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε την άποψη τη Επιτροπής και να δώσουμε ω μήνυμα προς την Επιτροπή Ανάπτυξης ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τι ευρωπαϊκά ταμεία χρειαζόμαστε και τι ευρωπαϊκά ταμεία χρησιμοποιούμε για το θέμα τη μετανάστευση. Το πλωτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ήγηρα για να εξηγήσει στον κόσμο, στον Ήγηρα, ότι δεν είναι παράδεισος η Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το χρηματοδοτούμε από τα ταμεία ανάπτυξης, αλλά και τα ταμεία που προέρχονται από τις ιστορικές υποθέσεις και χρησιμοποιούνται για τρίτες χώρες. Η συνεργασία για την ανάπτυξη έχει να κάνει με την ανάπτυξη, αλλά η μετανάστευση και η καταπολέμηση της μετανάστευσης, γιατί δυστυχώς εκεί το θέτουμε το θέμα, είναι ε, θέματα τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τους ίδιους πόρους τα ίδια κονδύλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λέει η Πρόεδρος, θα το έχουμε αυτό υπόψη όταν θα κοιτάξουμε και την γνωμοδότηση της ΔΕΒΑ. Ο κύριος Γκυρέος Σαλόμ και μετά ο κύριος Νόιζερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους ομιλητές Φαίνεται ο βασικό εχθρό που έχουμε εκεί για να εδραιώσουμε μια συνεκτική πολιτική και κοινή κυρίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καταπολέμηση της χειραγώγησης της κοινή γνώμη. Όπω είπε και ο κύριο Αμπρόση, εκεί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλοί μύθοι που κυκλοφορούν για τη μετανάστευση και θα ήθελα να προσθέσω και εγώ μερικού. Αν δούμε τα πραγματικά στοιχεία, το ισοζύγιο της κλασικής μετανάστευσης δεν έχει αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Αυτό που έχει αυξηθεί είναι η πίεση που προέρχεται και που παράγουν οι εμπόλεμες σειράξεις και οι ανθρωπιστικές κρίσεις που απορρέουν. Λέγουν στους πολίτες ότι έχουμε χιονοστιβάδα τέτοιων μεταναστών τώρα. Αν όμως κοιτάξουμε τα στοιχεία, παρά τα όσα είπε και η κυρία Βίξτρομ και η κυρία Σλάιν, ότι κάποιες χώρες δέχονται περισσότερες από, ε, από κάποιες άλλες, είναι γεγονός ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδεχόταν όλους τους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες όπως ο Λίβανος ε, αναλογικά θα είχαμε 8 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Ισπανία και 20 εκατομμύρια στη Γερμανία. Καμία λοιπόν χιονοστιβάδα. Κοινωνικές υπηρεσίες. Ήθιστε να λέγεται ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες καταραίουν γιατί έχουν κατακλειστεί από τους μετανάστες. Ποιο είναι το γεγονός. Δείχνουν όλες οι μελέτες ότι η μετανάστευση συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και για λόγους δημογραφικούς και ηλικία κοστίζει περισσότερη μετανάστευση από ό,τι αποφέρει. Ασφάλεια τώρα. Έχουμε δει όλοι ότι οι περιπτώσεις μειωμένης ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους τελευταίους μήνες δεν γίνονται από μετανάστες αλλά ανθρώπους που έχουν γεννηθεί, μορφωθεί, μεγαλώσει στη χώρα όπου έγινε το εκάστοτε συμβάν και η παραβίαση της ασφάλειας. Μέγα λοιπόν το έργο που έχουμε μπροστά μας να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, τη χειραγώγηση της κοινή νόμης και ίσως έχει έρθει η ώρα, όπως είπε και ο Κόνι Ρόιτερ, να ακούσουμε το άλλο τραγούδι του Μάνο Τσάου, επόμενο σταθμό η Ελπίδα, πρόξιμα στασιόν Περάσα. Um, Ευχαριστώ κύριο Νόιζερ και μετά ο κύριο Μανσκούρ, τελευταία ομιλητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να θέσω ερωτήσεις, μάλλον να απευθύνω μια έκκληση σε εμάς τους ίδιους. Νομίζω ότι έχουμε επαρκώς να περιγράψει την κατάσταση. Έχουμε αναλύσει τη διάθεσή μα. Θα πρέπει να δούμε πώ ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω βουλευτέ, μπορούμε να δράσουμε πλέον. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Έτο Ανάπτυξη θεωρώ ότι έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να δράξουμε για το λόμπι για τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη, για μεγαλύτερη συνεργασία για την ανάπτυξη, να ενισχυθούν όλα αυτά. Τα τελευταία χρόνια η εργασία αυτή, ε, το λόμπι αυτό έχει πληχθεί τα πλούσια κράτη είχαν υποσχεθεί 0,7% του προπολογισμού τους για αναπτυξιακή συνεργασία. Εγώ είμαι από μια πλούσια χώρα και αυτή η πλούσια χώρα τις 15, τα τελευταία 15 χρόνια ε, είχε σοσιαλιστικές, ε, δεξιές, ε, κυβερνήσεις, κυβερνήσεις από όλο το πολιτικό φάσμα αλλά δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε στο θέμα της χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Και είμαστε στο επονίδι στο 0,4% κάπου στη μέση. Λίγο παραπάνω από αυτά που ζητάμε από τις ε, καινούργιες χώρες της ε, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι στο 0,33%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της χρηματοδότησης και θεωρώ ότι τη διάσκεψη του Ιουλίου στην Αντίσα Μπέμπα θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε προκειμένου να παρουσιάσουμε μια κοινή τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη. Να υπάρξει μια επιτέλου μεγαλύτερη κίνηση. Ο Μέρκελ και ο Λάντ ε, συνασπίστηκαν και υποστήριξαν ο ένα τον άλλον για το θέμα τη Ουκρανία. Αυτό το εκτίμησα. Θα ήθελα λοιπόν συμβολική τέτοια δράση, αλληλεγγύη και για την αναπτυξιακή συνεργασία. Thank you, Mr. Mansko, and then Mr. Leeds has sneaked in the last minute. So, Mr. Mansko, then Arne Leeds, and that's the last. Κύριος Μανσκούρ, εγώ θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τους ε, εισηγητές που παρενέβησαν και τον ανθρωπιστικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη μετανάστευση από αρχαιοτά των χρόνων οι άνθρωποι πάντοτε μετακινούνταν. Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα. Όμως ε, σήμερα τίθεται το εξής ερώτημα. Υπάρχει πρόβλημα για τη μετανάστευση. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μετανάστευση, την δομούμε, την σκεφτόμαστε, τη δίνουμε ένα κοινωνικό, νομικό και ανθρωπιστικό πλαίσιο και αυτό θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τον κόσμο να μετακινείται. Όταν έχουμε να κάνουμε με φόβο, δικτατορία, πείνα, ανησυχία και βλέπουμε τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, ε, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τον κόσμο να έρχεται εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το νομικό πλαίσιο, γιατί ακόμα και αν δεν το κάνουμε τώρα, ε, θα ξανάρθουν ε, και δεν τους αφήσουμε να έρθουν με ανοιχτή πόρτα από την μπροστινή πόρτα, θα έρθουν από την πίσω πόρτα γιατί θα φοβούνται πάντοτε οι άνθρωποι. Και αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι τι θα κάνουμε όταν θα έρθουν, να τους δεχτούμε με τρόπο καλό, να μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα, ένα αρμονικό πλαίσιο. Αυτό επιθυμούμε. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα μετανάστευσης, εμείς έχουμε το πρόβλημα του πώς θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα αντιληφθούμε το θέμα της μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομος θα είμαι. Σε σχέση με αυτά που είπε ο Νόρμπερτ Νόιζερ, πολύ σύντομα μια δήλωση από πλευρά μου. Εμείς πώς μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε ως βουλευτές. Φέτος στη Γερμανία θα φιλοξενήσουμε τη Σύνοδο Κορυφής των G7 με θέμα βασικό την Αφρική. Εδώ και μια εβδομάδα με προβληματίζει. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε το ενακτήριο λάκτισμα εκεί. Ε, αξιοπρεπής δουλειά παγκοσμίω ήταν το σύνθημα των συνδικάτων που είχαν μια διάσκεψη στη Γερμανία. Κάναμε και κοινή ακρόαση για την αξιοπρεπή εργασία με το ΕΛΚ και αυτό θα πρέπει να ε, τονίσουμε. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αποφασίσουν κάτι σχετικά τις επόμενες εβδομάδες, να το υποστηρίξουμε και να το εγγράψουμε στην ημερήσια διάταξη και να καλέσουμε τη Σύνοδο Κορυφής του G7 να αναλάβει περισσότερες δραστηριότητες και στα πλαίσια του έτους της ανάπτυξης. Μια ιδέα για τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Um, πολύ ωραία ιδέα. Για το G8. Giving the chair uh, Πριν ξαναδώσω τώρα την Προεδρία στην κυρία Γκάλ Πέλτς, είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και έχουν τίποτα να προσθέσουν. Um, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, γι' αυτό λοιπόν ε, θα μιλήσω επιγραμματικά. Το θέμα αυτό παραμένει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας και των πολιτικών προτεραιοτήτων, αποτελεί άλλο το τμήμα και των κατευθυντηρίων γραμμών του Πρόεδρου Γιούγκερ. Στο πλαίσιο αυτό, όταν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τον ε, αναπτυξιακό αντίκτυπο της μετανάστευσης, αυτό θα παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα και θα δώσω το λόγο και στον συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση και όχι μόνο για τη διεθνή συντεύκο δηλαδή. Δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε αυτό μόνο από γραφειοκρατική άποψη. Για κάποιου ανθρώπου αυτό αποτελεί με το μοναδικό τρόπο πραγματικά να επιβιώσουν. Η μετανάστευση δεν αποτελεί κατά βάση αποτυχία τη ανάπτυξη. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το βιωτικό επίπεδο της χώρου του Νότου εν γέννη, αλλά αυτό μπορεί να αυξήσει και όλα τις ε, μεταναστευτικές ροές, γιατί ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα και τα μέσα για να μεταναστεύσει, που δεν είχε ενδεχομένω στο παρελθόν. Να το έχουμε λοιπόν αυτό την υπόψη. Επίσης, ότι οι μετανάστες ε, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στη χώρα προέλευσης και στη χώρα υποδοχής. Ένας βουλευτής μίλησε για τον όγκο των εμβασμάτων. Τετραπλάσιο ποσό, τετραπλάσιος όγκος από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σήμερα. Δεν μιλάμε για μικρό ποσά. Πολύ πιο πολλά από αυτά που δημόσια χορηγούμε. Ο ρόλος της αναπτυξιακής συνεργασίας για τη μετανάστευση διτός, εν συντομία, να βελτιώσουμε τους κανόνες για τη μετανάστευση για να είναι πιο αποτελεσματικοί και νομίζω ότι αυτό προτάθηκε ως ιδέα εδώ στη συζήτηση και κατά δεύτερον θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα της ε, άτυπης μετανάστευσης. Της παράτυπης μετανάστευσης. Αναφέρθηκε και η διακίνηση των ανθρώπων. Σίγουρα πρόκειται για κάτι το οποίο καταπολεμούμε. Πολλά θα είχα να πω ακόμη. Λυπάμαι που χρειάστηκε να είμαι τόσο σύντομο. Αν θα επιτρέψετε, ο συνάδελφο ε, θα ήθελε να σα διώξει και την ιστορική διάσταση από την Γενική Διεύθυνση Home. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζουμε την ανάγκη να υπάρχει πραγματικά κοινή συνεδρίαση μεταξύ των Επιτροπών εδώ στο Κοινοβούλιο για να υπάρχει συνοχή στο Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί μάλιστα και αυτή την ίδια προσέγγιση. Επί σειρά ετών η DG Home και η DG DEFCO ε, συνεργάζονται εντονότατα και προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη στη μετανάστευση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Δεν έχουμε και χρόνο άλλωστε. Και άλλωστε και ο συνάδελφος έχει πει πολλά βασικά. Θα ήθελα να αναφέρω την ατζέντα για τη μετανάστευση που περιμένουμε ότι θα έχει εγκριθεί μέχρι τέλη Μαΐου. Όπως είπαν πολλοί, η μετανάστευση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προαπαιτεί συνεκτική και μακροπρόθεσμη πολιτική αντίδραση. Σήμερα δεν μίλησα για ολιστική, συντολική προσέγγιση. Θα μπορούσα να το έχω κάνει, με το έκανα όμω. Γιατί. Θα πρέπει παρόλα αυτά να υπάρχει συνολική προσέγγιση. Η ατζέντα θα οικοδομηθεί, θα στελεχωθεί βάσει των προτεραιοτήτων του Πρόεδρου Γιούγκερ. Αποτελεσματική πολιτική για την άσυλο, καταπολέμηση της άτυπης, παράτυπης μετανάστευση και η εξωτερική διάσταση της διασφάλισης και της ε, προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Σκοπός είναι η ατζέντα να εξετάσει όλη τη διαδικασία από τη χώρα προέλευσης, μέσω της χώρας διέλευσης, μέχρι τη χώρα υποδοχής στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και το πώς ε, γίνεται η υποδοχή των μεταναστών εκεί. Να αναφερθώ επίση στο εξή. Η αναπτύξη αναπτύξιακή συνεργασία θα αναφερθεί αυτό και στην ε, ατζέντα. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τις χώρες εταίρες. Για να τονίσουμε τα κρυφά αίτια της μετανάστευσης και να επωφεληθούμε και από τις ευκαιρίες της μετανάστευσης. Μιλήσαμε πάρα πολύ σήμερα για τους κινδύνους, για τα τραγικά περιστατικά στη Μεσόγειο όπου χάνει ο κόσμος τη ζωή του. Αλλά υπάρχουν και ευκαιρίες που θα πρέπει να δράξουμε. Δεν υπάρχουν μόνο ρίσκα και κίνδυνοι. Θα πρέπει να επωφεληθούμε, να μεγιστοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες και για την χώρα προέλευσης και για τη χώρα υποδοχής και στην Ευρώπη και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σας ευχαριστώ. Thank you very much for the commission. Thanks for the... Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστούμε και για τις παρεμβάσεις. Τώρα έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και πραγματικά είναι μεγάλο, μεγάλη πρόκληση. Τέσσερις ομιλητές, πέντε λεπτά ο καθένας για να απαντήσετε στα θέματα αυτά. Πιο λίγο, πιο λίγο λέει η πρόεδρος. 35 maximum. Okay, 35 maximum. So, uh, we have to finish at 35. Να κλείσουμε στις 12 και 35. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Αμπρόζη και να ακολουθήσουμε τη σειρά των ομιλητών. Brief as possible. Ευχαριστώ. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Thank you. Η εξωτερήκευση, το outsourcing δεν είναι κάτι που εγώ θα υποστήριζα. Τώρα όσον αφορά την διάσωση ζώων, οποιοδήποτε είδος συνεργασίας είναι πρόσδεκτο. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά από τη διάσωση. Ε, τι γίνεται με την ε, την βοήθεια που δίνεται μετά. Τι συμβαίνει μετά σε αυτούς όταν διασωθούν και βγουν στην στεριά. Στο παρελθόν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εξωτερικεύσει τον ε, συνοριακό έλεγχο, ιδιαίτερα με το προηγούμενο καθεστώς της Λιβύης, αλλά δεν θέλουμε καθόλου να φτάσουμε στο ίδιο μοντέλο. Η προτεραιότητα θα είναι και θα πρέπει να είναι η προστασία των ανθρώπων και όχι μόνο η προστασία των συνόρων. Δηλαδή η προστασία των συνόρων μέσω της προστασίας των ανθρώπων και όχι αντιστρόφως. Υπάρχει επίσης το θέμα της αξιοπιστίας όταν μιλάμε για την εξωτερήκευση του ε, ασύλου. Ακούσαμε και ότι ένα από τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εσωτερική αλληλεγγύη, δηλαδή ε, η μοιρασιά του βάρους ανάμεσα στους 28. Και είναι κάπως παράξενο να ζητάμε από άλλες χώρες εκτός, την Ευρώπη, Ευρώπης να δείξουν ε, αλληλεγγύη και ε, να μοιραστούν το βάρος, ενώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχουμε ακόμα αυτό καταφέρει. Είναι θέμα αξιοπιστίας Τη της Ένωσης νομίζω που θέλει να είναι ένας παγκόσμιος παίκτη και όχι απλά ένας παγκόσμιος πληρωτής, όπως έχει υποθεί για το θέμα των ποσοστώσεων. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να εξασφαλίσει τα 28 κράτη-μέλη έχουν ε, την ίδια, το ίδιο ενδιαφέρον για τη διαχείριση της εισρωής, της μετανάστευσης. Ε, θα πρέπει να δούμε και να κάνουμε ότι είναι λογικό και αποδεκτό. Κάτι τέτοιο θα ήταν μια μεγάλη βελτίωση. Πιστεύω πως είναι σημαντικό η πρόταση αυτή των ανθρωπιστικών διαδρόμων είναι αλήθεια ότι ε, θα ενοχλούσε το επιχειρησιακό μοντέλο των διακινητών και των λαθρεμπόρων δεν θα πρέπει όμως να πιστεύουμε πως τα προβλήματα συμβαίνουν αλλού ε, και στην Ευρώπη υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή το δίκτυο δεν είναι ανεπαρκές. Η σοβαρή όμως αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου θα πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Και η αρχή την οποία εμείς υποστηρίζουμε, το μοντέλο που υποστηρίζουμε, ε, το κάνουμε γενικώ και όχι μόνο για εδώ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, ε, ε, νομίζω πως αυτό γίνεται πολύ καλά. Στην Τουρκία, σε μια εβδομάδα, μπήκαν τόσοι πρόσφυγες από τη Συρία όσοι στην Ευρώπη ένα ολόκληρο χρόνο. Κέρας της Αφρικής. Εκατομμύρια πρόσφυγες στα στρατόπεδα και προσφύγων εδώ και 20 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πως, ποιο είναι το μοντέλο στον κόσμο Ακούσαμε το μοντέλο της Αργεντινής, ε, διακυβέρνηση της μετανάστευσης, αυτό είναι ένα μοντέλο που θα πρέπει να μελετήσουμε. Ευχαριστώ, ο ε, Πρέζης Φραμντέο. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιες παρατηρήσεις και σχόλια για το θέμα της επεξεργασίας ε, των αιτήσεων των ετών των άσυλων και των προσφύγων σε τρίτες χώρες, την, την εξωτερική ε, ανάθεση των επιχειρήσεων διάσωσης, η Αφρικανική Ένωση δεν έχει συζητήσει αυτή τη δυνατότητα. Ωστόσο, θα ανέμενε κανείς ότι η απόφαση θα ήταν να το αποθαρρύνουμε ε, όσο γίνεται περισσότερο, γιατί θα θεωρείται σαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ποσεί τις ευθύνες της όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών. Επίσης, θα μοιραζόμασταν ε, την, ε, τον έλεγχο και τη διαχείριση της μετανάστευσης ε, στην επικράτεια της Ένωσης. Από την άποψη, λοιπόν, της Αφρικανικής Ένωσης θα αποθαρρύναμε αυτή την ε, εξωτερική ανάθεση. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ποια είναι η πολιτική της γειτονίας. Έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Ποιος παρακολουθεί την διαδικασίες που θα δημιουργηθούν τις, τις, τις δυνατότητες, ποιος εκπαιδεύει το προσωπικό που κάνει αυτή τη δουλειά και τέλος ποιος είναι υπόλογος, ποιος είναι υπεύθυνο. Δεν μπορεί κανείς να πληρώνει για υπηρεσίες απλά και να παραδίδει έτσι την ευθύνη σε κάποιον άλλον για τέτοια σημαντικά θέματα. Το θέμα τώρα το εκπαιδευτικό. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό η εκπαίδευση να γίνεται και από τις δύο πλευρές, και από την Αθήνα και από την Ανατολή και από την Ασία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η ολοκλήρωση σε κοινοτικό επίπεδο. Να υπάρχει δηλαδή αποδοχή ώστε να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε κάποιους τομείς της κοινότητας της μεταναστευτικής από το να αισθάνεται αποκλεισμένη και να προβαίνει έτσι σε δράσεις οι οποίες είναι καταδικαστές. Τώρα, η χιονοστιβάδα μεταναστών για τους οποίους μιλάμε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δεχτούμε το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις Αυτές οι κρίσεις έχουν ε, εκραγεί και είναι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Οι Σύριοι ποτέ δεν επέλεξαν να πέσουν σε κρίση, ούτε οι Ιρακινοί ούτε οι Λιβύοι. Ποιος ευθύνεται λοιπόν για αυτήν την κατάσταση? Ας μην αρνούμαστε ότι υπάρχει κοινή ευθύνη για την ανθρωπιστική κρίση όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Πρέπει γι' αυτό το πράγμα να είμαστε έντιμοι. Και επίσης, κάποια στοιχεία. Τα εμβάσματα για τα οποία μιλάμε είναι συν πλήν 60 δις ετησίως που πάνε στην Αφρική. Οι παράνομες οικονομικές ροές από την Αφρική όμως είναι πάνω κάτω 50 δις. Τώρα, αν αυτά τα χρήματα μπορούσαν να μπουν σε κοινή ανάπτυξη, ε, ε, ε, θα, γινόταν, θα υπήρχε πολλή ανάπτυξη. Η έκκληση είναι ας κάνουμε αυτό που είναι σωστό. Θα ήταν πραγματικά ανήθικο και ασυνείδητο το να κλείνουμε τα μάτια και να μην τοποθετούμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο στην μετανάστευση. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη, κύριε Παπαδοπούλου. Δεν μπορώ να αντισταθώ να κάνω πρώτο σχόλιο. Οι περισσότερε ερωτήσει ε, και αντιδράσει ήταν για την πρόσβαση στην Ευρώπη και την κατάσταση στην Ευρώπη σε μια συζήτηση που, ο, τίτλο είναι Ανάπτυξη και μεταναστε... Ε, βοήθεια και μετανάστευση. Αν σκεφτούμε τα παιδιά που είναι πρόσφυγες στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Πώς, ε, τι μπορούν να κάνουν ο Λίβανος και η Ιορδανία, για πόσο καιρό. Εάν δεν το σκεφτούμε αυτό, απλά μιλάμε για συμπτώματα και μιλάμε για τις αφήξεις στην Ευρώπη μόνο. Τα δύο θέματα για την ε, εξωτερική ανάθεση και το σύστημα των ποσοστώσεων. Πολλά υπόθηκαν ήδη για την ε, εξωτερική ανάθεση και ανησυχίες υπάρχουν, ιδιαίτερα ε, τα τελευταία λόγια του πρέσβη δεν είναι νέα αντίληψη αυτή, δεν, ήδη από το 2003 έχει συζητηθεί και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ευθύνη αυτών των ανθρώπων, για αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν σε διάφορα μέρη ε, εκτός της Ευρώπης. Τι γίνεται με όλους αυτούς. Μπορεί να περιμένουν για ένα χρόνο, για δύο. Τι γίνεται εκεί, ποιος είναι υπεύθυνος. Έχουν, έχουν πρόσβαση σε νομική βοήθεια, έχουν τα δικαιώματα και τις εγγύσεις που θα έπρεπε να έχουν όταν εξετάζονται οι αιτήσει τους. Μπορούν να ζητήσουν άσυλο ε, στην Ευρώπη και βέβαια ποτέ δεν θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ε, ε, προηγούμενης της προηγούμενης τους προέλευσης. Δηλαδή, και όταν πρόκειται για αυτά που ανέφερε η Σεσίλια Βέξτρομ. Γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι η ποσόστοση για επανεγκατάσταση, που είναι κάτι διαφορετικό και ένα πιθανό σύστημα ποσοστώσεων για του ετούντε άσυλου που φτάνουν διαρκώ. Είναι κάτι το άλλο. Είναι δύο χωριστά πράγματα. Ποσοστώσει που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με την έννοια ότι θα γίνουν κοινέ ευρωπαϊκέ προσπάθειε για, ε, για κάποια ρύθμιση αυτό είναι κάτι που πιστεύω έχει υποστηριχθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ανάγκη να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης αλλά όταν πρόκειται για τους ετούντες άσυλο είναι κάπως πιο περίπλοκα τα πράγματα ε, και η Sky Keller το ανέφερε αυτό. Έχουμε οικογενειακούς δεσμούς, θα έχουμε πάντοτε ανθρώπους που θέλουν να πάνε αλλού, ακόμα και αν έχουμε ορισμένα νούμερα από τα κράτη-μέλη Και μετά έχουμε διαφορετικές δυνατότητες ε, ε, ένταξης και υποδοχής στα κρατημέλη. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό, δεν υπάρχει τρόπος να υποδείσει τον κόσμο να γυρίζει γύρω-γύρω. Και εκτός αν δεν έχει ένα ε, επίπεδο αλληλεγγύης, δεν θα μπορείς να αντιμετωπίσεις το θέμα ότι ο κόσμος όλος αυτός θα κινείται στα διάφορα Ευχαριστώ. Κύριο Σρόιτερ. Σας ευχαριστώ πολλά. Ακούσαμε για το σύστημα το ποσοστώσεις και για το θέμα του outsourcing της εξωτερικής ανάθεσης. Φανταστική η εξωτερική ανάθεση και κοιτώντας τι έχουν κάνει οι Αμερικανοί με την εξωτερική ανάθεση του πολέμου σε ε, εταιρείε και βλέπουμε ότι έχουμε κέντρα τα οποία στην Ευρώπη τα διαχειρίζονται εταιρείε. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να διδοκοποιηθεί ο τομέα αυτό και αυτό με φέρνει σε ένα άλλο θέμα. Μιλάμε για τα 0,7% για αναπτυξιακά ζητήματα. Δεν μιλήσαμε όμω για ένα συγκεκριμένο θέμα, η ανάπτυξη δυναμικού capacity building, εντετέρως για την κοινωνία, του την κοινωνία των πολιτών, για τι δύο πλευρέ τη Μεσογείου. Γιατί αυτό τι σημαίνει, σημαίνει παιδεία, σημαίνει όχι μόνο το επίσημο σχολικό σύστημα, αλλά και ελεύθερος χρόνος ε, πολιτισμός, ε, κουλτούρα, πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, πώς να τις πω, δραστηριότητες. Αυτό είναι ανάπτυξη δυναμικού. Δυναμικό επίσης για τις ΜΚΟ. Ένα μέλος από την Νορβηγία. Καθάρισαν τα σύνορα μεταξύ Ιορδανίας και Συρίας. Έχουν αφαιρέσει στα τελευταία χρόνια 50.000 νάρκες. Αυτό είναι ανάπτυξη δυνατοτήτων. Σημαίνει δηλαδή δυνατότητα να δράει κανείς, να κανείς στα καταλήμματα προσφυγικά, στην Ιορδανία, στο Λίβανο. Αυτό τι σημαίνει. Αναγνώριση του ρόλου και της ανάγκης δράσης. Θα επανέλθουμε στο θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δούμε σε ποιον απευθύνονται τα χρήματα. Όταν μιλάμε λοιπόν για συνόδους, όπως έκανε η συνάδελφος, καλό είναι αυτό να τεθεί στο θέμα της σημερινής διαταξή και εν ώψη των συνεδρίων, αλλά να συνδέεται και με άλλα θέματα κοινωνικής προστασίας. Θα πρέπει να ειδωθεί υπό την έννοια της συνεργασίας Οι πάροχοι ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν και αυτοί οι συνδικάτα, αλλά οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, γενικά έχουν καλή φήμη γιατί ξέρουν πώς ε, δρούν αποτελεσματικά και είναι καλέ στο έργο του. Άρα η σύνοδο είναι πάντα καλή για την πολιτική ευαισθητοποίηση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν καλά στοιχεία. τέλο. δεν μπορώ να αποδεχτώ το θέμα του, του λαθρέου. Δεν υπάρχει τίποτα το λαθρέο, υπάρχει το παράτυπο μόνο αλλά θα έπρεπε να συμφωνήσουμε το θέμα, στο θέμα της ρολογίας. Ίσως και θα πρέπει και οι μεταφραστές να χρησιμοποιούν το παράτυπο μόνο και όχι το λαθρέο, το παράνομο. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά κατάλληλος ο όρος λαθρέος, παράνομος και θα σταματήσω εδώ, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για το ευρωπαϊκό έτος. Ανάπτυξης. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα του όρου, αλλά ασφαλώς οι διερμηνείς πάντα μεταφράζουν αυτά που λέει ο κόσμος. Ευγενικά ευχαριστεί η Πρόεδρος του Συρμηνής που έμεινε λίγο παραπάνω. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ καταρτίζει έκθεση. Εμείς θα γνωμοδοτήσουμε το θέμα αυτό. Ένα από τα πρώην αφεντικά μου μας είπε ότι έχουμε τρεις στίβες χαρτιών πάντα στο γραφείο μας. Ε, αυτά που μπαίνουν, αυτά που βγαίνουν και αυτά που ποτέ δεν μπορούν να φύγουν γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό λοιπόν το θέμα αποτελεί ένα από αυτά τα πολύ δύσκολα ζητήματα. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Ευχαριστούμε τους ομιλητές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήλθατε και μας μιλήσατε εδώ σήμερα το πρωί.